Λοιπόν, ξεκινούμε τη συνεδρίασή μας ή μάλλον συνεχίζουμε την πρωινή συνεδρίαση. Καλό απόγευμα σε όλους. Το πρώτο θέμα της ημέρησης διάταξης είναι αυτό που μας δίνει τη χαρά να υποδεχθούμε την ε, Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου για να μας παρουσιάσει το πρόγραμμά σας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου τη ελληνική Προεδρίας. Είχα την ευκαιρία να σα συναντήσω στην Ελλάδα στο ταξίδι της αντιπροσωπείας μας. Ήταν μια, ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι και είχαμε πολύ καλή υποδοχή από τη δική σας πλευρά και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ξέρω ότι έχετε πολλή εργασία να κάνετε αυτό το διάστημα. Όλες οι προεδρίες πρέπει να εργαστούν πολύ σκληρά με έναν τρόπο που είναι συγχρόνος και πραγματιστικός και με συμβιβαστικές λύσεις που πρέπει να δώσετε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη εποχή για όλες τις προεδρίες, αλλά φυσικά είναι και συναρπαστική. Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το, για το πρόγραμμά σας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Κυρία Κόλια, λοιπόν, σας χαιρετίζουμε θερμά και χαιρόμαστε που έχετε έλθει ενώπιον μας για να λάβετε το λόγο ενώπιον της Επιτροπής μας και ελπίζουμε ότι μπορούν να ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις μετά από την παρέμβασή σας, αλλά έχετε το λόγο καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω και πιστεύω ότι η ελληνική προεδρία σε ό,τι τουλάχιστον αφορά στο τομέα της ισότητας των φίλων, θα κάνει τα καλύτερα για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα, το δικό της ίχνος σε αυτόν τον αγώνα που καταβάλλετε εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα ίσα δικαιώματα γυναικών και ανδρών. Και για να περάσω την ομιλία μου. Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του Νότου βιώνουμε ακόμη και σήμερα τις φοδρές επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης. Ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει. Οι προβλέψεις της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωζώνη, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, περιγράφουν ένα μέλλον καθόλου εφησυχαστικό. Τοποθετούν το βιωτικό επίπεδο στον ορίζοντα του 2023 σε επίπεδα με τα βία συγκρίσιμα με Κίνα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1960. Αυτό, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι και το πλαίσιο της δικής μας δράσης κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Καλούμαστε ως Προεδρία να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων ενώ μεγάλα τμήματα της κοινωνίας μας υποφέρουν από την ανεργία τη φτώχεια και την περιθωριοποίηση. μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει πώς μπορεί να μιλάει κανείς για την ισότητα των φύλων όταν κάποιοι ευρωπαίοι συμπολίτε μας αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης. μήπως τελικά είναι μια πολυτέλεια για τις κοινωνίες μας. πρέπει να αντισταθούμε στην ευκολία αυτής της συλλογιστικής όχι μόνο γιατί αφορά τα δικαιώματα του μισού και πλέον πληθυσμού του πλανήτη μας, όχι μόνο γιατί η διασφάλιση της ισότητας των φύλων είναι θέμα δημοκρατίας, αλλά γιατί τελικά η ισόρροπη και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγή γνώσης, αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί μονόδρομο για την ευημερία των κοινωνιών μας. Η κρίση μέσα στα τόσα κακά που επέφερε μας έκανε να κοιτάξουμε και λίγο πίσω. Μας όθησε να ξανακοιτάξουμε κάποια νούμερα τα οποία ήδη ήταν γνωστά σε πολλούς από εμά. Αλλά περιέργως τα νούμερα αυτά δεν είχαν καταφέρει να σπάσουν τη γυάλινη οροφή του δημοσίου συμφέροντος. Η εξίσωση είναι απλή. Περισσότερες γυναίκες στην απασχόληση ισούται με μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα. Κατά τον ΟΟΣΑ, από το 1995 έως σήμερα, το ίμιση της αύξησης του ρυθμού απασχόλησης στην Ευρώπη και το 1 τέταρτο της οικονομικής ανάπτυξης οφείλονται στη μείωση του χάσματος μεταξύ ανδρικής και γυναικείας απασχόλησης. Για να περάσουμε από την άλλη πλευρά του πλανήτη, στην Ιαπωνία, η αύξηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό μετρίασε την αναπτυξιακή στασιμότητα και προφύλαξε την οικονομία της χώρας από μια βαθύτερη κρίση. Στη Λατινική Αμερική, επίσης οι εργαζόμενες γυναίκες βοήθησαν να μειωθεί η φτώχεια για οικογένειες με δύο γονείς από το 40% στο 26% κατά τη διάρκεια του 2007 Όμω κάποιο θα μπορούσε να διατυπώσει και αντιστρόφως το ζήτημα που μα απασχολεί. Θα μπορούσε να μα πει ότι η ανισότητα των φίλων κοστίζει τελικά. Κοστίζει οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Για παράδειγμα, η ανισότητα πρόσβαση στην αγορά εργασία έχει αυτό κόστο ευκαιρία. Το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο εργάζεται μόλι το μισό ενεργό εργατικό δυναμικό γένου θηλυκού αυτό κυρίε και κύριοι συνεπάγεται χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με το διεθνές νομισματικό ταμείο έως και κατά 27% του αεπ. για να γυρίσω τώρα λίγο στην ευρώπη στην ήπειρό μας σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής επιτροπής εάν οι γυναίκες της ευρώπης απασχολούνταν στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας εξίσου με τους άνδρες το ευρωπαϊκό αεπ θα αυξανόταν ετησίως κατά 9 δισεκατομμύρια ευρώ εδώ να θυμίσω ότι αυτό ισοδυναμεί με 1,3 φορές το ΕΠ μιας χώρας, μιας μικρής χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή είναι η Μάλτα. Ακόμη μικρό μερίδιο γυναικών στην απασχόληση, κυρίε και κύριοι, σημαίνει μειωμένη οικονομική ανεξαρτησία και περιορισμένη συμμετοχή στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Η σημασία αυτή τη παρατήρηση αναδεικνύεται εάν σκεφτούμε ότι οι γυναίκε σήμερα ελέγχουν περίπου 23 δολάρια 23 δολάρια, επαναλαμβάνω, της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης παγκοσμίω. Κι όμως, μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ίμιση του πληθυσμού ως εξειδικευμένο κοινό. Βέβαια δεν σταματάμε εκεί, γιατί κόστος χαμένων ευκαιριών ανακαλύπτουμε και στα οικονομικά, πολιτικά και επιστημονικά κέντρα λήψη αποφάσεων. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η συμμετοχή των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων συνδέεται με αυξημένη κερδοφορία, μακροπρόθεσμη στοχοθεσία και μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους. Εταιρείε με διοικητικά συμβούλια που αποτελούνταν τουλάχιστον κατά το 1 τρίτο από γυναίκε δείχνουν κέρδη αυξημένα κατά 42%. Στους δε μετόχους φτάνουν μερίσματα αυξημένα κατά 53%. Παρ' αυτά, μόνο το 11% των γυναικών συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, ενώ λιγότερο από τα 3% αυτών των εταιριών διευθύνονται από γυναίκες. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμά τους αριθμούς που καταδεικνύουν τη χαμηλή συμμετοχή γυναικών τόσο στα όργανα λήψη αποφάσεων, τόσο οικονομικών όσο και πολιτικών, αλλά και στα πεδία της γνώσης και της επιστήμης αν υπάρχει κάποιο στοιχείο πολυτέλειας στην ισότητα των φύλων είναι η αντιμετώπιση της ως αξίας εντός εισαγωγικών πλην όμως ανεφάρμοστη στην πράξη. δεν μπορεί η ισότητα των φύλων τον 21ο αιώνα να συνεχίζει να αντιμετωπίζεται αφιψηλού μπροστά στο τεράστιο κοινωνικό κόστος που επιφέρει το έλλειμμά της. Απ' την άλλη όμως κυρίες και κύριοι παρατηρούμε ότι παρά το κόστος της ανισότητας των φύλων που όλοι αναγνωρίζουμε η κρίση ως σήμερα δεν έχει μετατραπεί τελικά σε ευκαιρία ενώ ο γυναικείο πληθυσμός ειδικά του ευρωπαϊκού νότου συνεχίζει να πλήττεται δυσανάλογα από την ύφεση διαπιστώνουμε συνεχώς τάσεις οπισθοδρόμησης. και τι εννοώ. οι γυναίκες πρωταγωνιστούν στην ανεργία στις κατώτερες θέσεις εργασιακής ιεραρχίας στις πρόσκαιρες και επισφαλείς μορφές απασχόλησης. τα ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας παραμένουν σταθερά χαμηλότερα από εκείνα των ανδρών με βάση τους δείκτες του 2012 όπως καταγράφονται στο κοινό πλαίσιο αξιολόγησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020 το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες ήταν μόνο 62,4% ενώ για τους άντρες 74,6%. Ιδιαίτερα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά και των μακροχρόνια ανέργων γυναικών. Και ενώ από την άλλη μέχρι το 2020 η Ευρώπη θα πρέπει να επιτύχει ένα ποσοστό 75% για τον πληθυσμό 20-64 ετών, οι γυναίκες παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διευρυμένο χάσμα δεξιοτήτων. Συνεχίζουν να επιλέγουν, αν μου επιτρέπετε να πω, γυναικείες σπουδέ με μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης. Την ίδια στιγμή όμως βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας αλληπάλληλες μελέτες που προέρχονται από την αγορά, όπως ενδεικτικά θα αναφέρω τελευταίες μελέτες της Manpower ή της McKinsey, οι οποίες υπογραμμίζουν ότι πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν θέσεις σε ειδικεύσει κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα της Μαρκίζη, η μία στις δύο ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας. Ελλείψεις δεξιοτήτων παρατηρούνται σε τομείς της επιστήμης επίσης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών. Όμως ακριβώς αυτή είναι η τομής όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται είναι ενδεικτικό ότι στις χίλιες γυναίκες πτυχιούχους στην Ευρώπη μόνο 29% κατέχουν πτυχίο πληροφορικής και μόνο 4 τελικά θα απασχοληθούν στον τομέα των ICT. Έτσι, στον κρίσιμο για την ανάπτυξη τομέα των ICT προσφέρει εργασία σε 7 εκατομμύρια ανθρώπους, οι γυναίκες συμμετέχουν μόνο κατά 30%. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να αναρωτηθούμε τελικά κάτι το οποίο το έχω αναρωτηθεί πάρα πολλέ φορέ προσπαθώντα να κάνω τη δουλειά μου ποια είναι η στάση τη κοινωνία απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα. παρά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση παρά την υιοθέτηση φαινομενικά σύγχρονων τρόπων ζωή οι κοινωνίε μα συνεχίζουν να λειτουργούν με βάση μια αναχρονιστική ιεράρχηση των φύλων. Μια ιεράρχηση τόσο παλιά ίσω όσο η ανθρώπινη ιστορία που όμως έχει φτάσει πραγματικά στα ωριά της, που δημιουργεί αδιέξοδα και παθογένειες στις κοινωνίες μας. Η άνεργη γυναίκα και πάλι φαίνεται σε καλύτερη υποψήφια για να υπομειστεί εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του σπιτιού, της ευρύτερης οικογένειας και των μελών που χρήζουν ειδική υποστήριξη. Αναθεωρείται τελικά μονομερό στο κοινωνικό συμβόλαιο. Ζητούμε από τη γυναίκα την επιστροφή στην φυσική, αν μου επιτρέπετε να πω, για το φύλλο τη κατάσταση τη μη αμοιβόμενη και ηθικά μη αναγνωρισμένη εργασία αυτό ο αναγκαστικό αλτρούισμό καθυλώνει όμω τη γυναίκα σε έναν ρόλο χωρί προοπτική. Γιατί ποιο μπορεί τελικά να είναι το μέλλον μια γυναίκα που δεν συμμετέχει στην κοινωνία τη γνώση, πώ θα επιβιώσει όταν ο επιστημονικό και τεχνολογικό αλφαβητισμός αποτελούν αυτονόητη προπόθεση για να λειτουργήσει ω πολίτης, ως γονέας, ασθενής, ψηφοφόρο κοινωνικών. Υπάρχει όμω και ένα ακόμα λόγο για να προωθήσουμε άμεσα τι πολιτικέ ισότητε των φίλων όταν η ανισότητα των φύλων και αυτό το ζούμε έντονα πλέον στην ελλάδα συνοδεύεται από τη φτώχεια και την απομόνωση τότε το μείγμα γίνεται εκρηκτικό. απειλείται η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ειρήνη. Έχουμε ακόμα πιο έντονα φαινόμενα ακραίων πράξεων βίας ενάντια σε γυναίκες. Αυξάνεται το εμπόριο γυναικών, η κακοποίηση, η ψυχολογική και σωματική βία, η ενδοοικογενειακή βία και η Έχουμε έξαρση σε φαινόμενα πολλαπλών διακρίσεων και εννοώ τη ρατσιστική βία κατά των γυναικών ή και τον κοινωνικό στιγματισμό. Τώρα για να μην σας κουράζω άλλα με αυτή τη γενική τοποθέτηση θα ήθελα να περάσω στο κομμάτι της Προεδρίας, της ελληνικής Προεδρίας στο τομέα της ισότητας των φύλων. Βασιζόμενοι σε αυτά που σας ανέφερα πριν λίγο, με το πρόγραμμα δράσης της ελληνικής προεδρίας του συμβουλίου της ευρωπαϊκής ένωσης στο τομέα της ισότητας των φύλων επιδιώκουμε και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομικής συγκυρίας. Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην αναπτυξιακή στοχοθεσία του στρατηγικού κειμένου Ευρώπη 2020. Να προχωρήσουμε ακόμη ένα βήμα προς την ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας. Εδώ θα ήθελα να, να τονίσω ότι το πρόγραμμα δράσεων που θα ακούσετε στη συνέχεια έχει εμπλουτιστεί με προτεραιότητες που προήλθαν από την κοινωνία των πολιτών ύστερα από σχετικό διάλογο που κάναμε με τις γυναικείες οργανώσεις κατά τη διάρκεια του 2013. Ας ξεκινήσουμε από τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών οργάνων. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί καταρχάς θεωρούμε σημαντική η υποχρέωσή μας την ενημέρωση και το συντονισμό των ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών οργάνων με αρμοδιότητα στην ισότητα των φύλων. Έχουμε λοιπόν προγραμματίσει για τον επόμενο μήνα, τον μήνα Φεβρουάριο, την ενημέρωση των Επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τι πολιτικέ ισότητε των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, το ΕΓΕ. Σε επίπεδο τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνουμε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου συνάντηση στην Αθήνα της ομάδα υψηλού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις. Στη συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατικών φορέων ισότητας όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και το ΕΓΚΕ. Κεντρικός μας άξονας είναι οι γυναίκες και η οικονομία. Ο βασικός αυτός άξονας αποτελεί και το πρόγραμμα δράσης μας. Το θέμα μας, όπως σας είπα, είναι οι γυναίκες και η οικονομία. Μέσω αυτού του κεντρικού άξονα επιδιώκουμε να αναδείξουμε τομείς πολιτικής που συμβάλλουν στη θωράκιση των γυναικών της Ευρώπης ενάντια στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Γιατί είναι σαφές πλέον ότι η οικονομική κρίση, ήδη σας τον ανέφερα και λίγο πιο πάνω, έχει και γυναικείο πρόσωπο, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου. Και ίσως το γυναικείο πρόσωπο είναι ακόμα πιο έντονο και πιο δύσκολο στο επίκεντρο λοιπόν των πολιτικών πρωτοβουλειών μας έχουμε θέσει την προώθηση των οικονομικών δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας των γυναικών, την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και την επίτευξη κατάλληλων εργασιακών συνθήκων. Στο ίδιο επίκαιρο θέμα γυναίκα και οικονομία, επιλέξαμε να επικεντρωθεί και η αποτίμηση της προόδου από την εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του προγράμματος δράσης του Πεκίνου. Την μεγάλη εικόνα στο τομέα αυτό, στο τομέα της απασχόλησης των γυναικών στα κράτη-μέλη, θα μας δώσει μελέτη που εκπονεί το ΕΓΕ, η οποία θα παρουσιαστεί σε ανοιχτή εκδήλωση στην Αθήνα στις 6 και 7 Φεβρουαρίου. Επίσης σκοπεύουμε, και πρέπει να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φίλων της Ελλάδας, να εισαγάγουμε μια νέα δυναμική που θα φέρει πιο κοντά τις γυναίκες στις τεχνολογίες, πληροφορίες και επικοινωνίες και στην ψηφιακή οικονομία θέλουμε να στρέψουμε το γυναικείο ταλέντο που σήμερα μένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό στο τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Γιατί όπως αποδεικνύουν διαδοχικές μελέτες, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης ακόμη και σε αυτήν εδώ την εποχή, την εποχή της κρίσης. Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και τις γυναίκες, καταγράφεται ένα έλλειμμα δεξιοτήτων νέων τεχνολογιών που αντιστοιχεί σε 500.000 θέσεις εργασίες μέχρι και το 2015. Το 2015 να σας θυμίσω είναι σε δύο ακριβώς χρόνια ή ξεκινάει σε ένα χρόνο. Αυτά δεν είναι αποτελέσματα μιας οποιασδήποτε μελέτης. Αυτή η μελέτη έχει ολοκληρωθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ελλάδα ήδη αναπτύσσουμε μια ευρεία και πολυμετοχική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τίτλο Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναική Απασχόληση βασισμένη στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας η ψηφιακή συμμαχία ακολουθεί το πρότυπο της δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Grand Coalition for Digital Jobs. Δημιουργήθηκε έτσι ένα ισχυρό εταιρικό σχήμα 15 φορέων από το χωρό της απασχόλησης και της πληροφορικής που περιλαμβάνει τους ακόλουθους. Coordinator, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας και οι υπόλοιποι που δουλεύουμε μαζί είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, ο Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας. Από πλευράς πανεπιστημίων μέχρι στιγμή συμμετέχουν το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τον τομέα ηλεκτρικών βιομηχανικών διατάξεων και συστημάτων αποφάσεων του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο σύνδεσμος επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών ελλάδας η cisco systems ελλάς η google η manpower group greece η microsoft ελλάς η oracle ελλάς καθώς και ο τομέας γυναικών μάνατζερ και επιχειρηματιών της ελληνικής εταιρείας διοίκησης επιχειρήσεων. Στο εταιρικό σχήμα αυτό συμμετέχει και η ομάδα Ευρώπη, η γνωστή ω Team Europe, της τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη, την προώθηση και τη διάχυση τη πρωτοβουλία αυτή. Το σχήμα αυτό δεν είναι κάτι στατικό, είναι δυναμικό. Αυτή είναι μόνο η αρχή και ο σκοπός μας είναι να, να συμμετάσχουν ακόμα περισσότεροι δημόσιοι φορεί όσο και εκπρόσωποι τη αγορά. Σκοπός λοιπόν είναι στη βάση του πρωτοκόλου, ενός πρωτοκόλου συνεργασίας και με κοινό σχεδιασμό όλων αυτών των φορέων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι φορείς να συνεργαστούν για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων. Επιτυχάνουμε συνέργειες, αξιοποιούμε διαθέσιμους πόρους και τεχνογνωσία, λαμβάνοντας υπόψη καλές διεθνείς πρακτικές. Το πρόγραμμα της συνεργασίας περιλαμβάνει δράση ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, απασχόληση και επιχειρηματικότητας γυναικών και νέων, καθώ και δράσει κατά πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση στι της τεχνολογίε και τη ψηφιακή οικονομία. Την εμπειρία αυτή, την εμπειρία τη ελληνική ψηφιακή συμμαχία, θα επιδιώξουμε να μοιραστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να καλέσουμε σε συντονισμένες δράσεις υπέρ της διάδοσης των νέων τεχνολογιών στο γυναικείο πληθυσμό. Γι' αυτό το λόγο στις 4 Απριλίου διοργανώνουμε Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα γυναίκες και ψηφιακή απασχόληση σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες. Μια ακόμα δράση όμως για να τελειώσω με τις δράσεις που προγραμματίζουμε έχει να κάνει με την γυναική απασχόληση και ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για το λόγο αυτό στις 27 και 28 Φεβρουαρίου διοργανώνεται πάλι στην Αθήνα συνάντηση διαβούλευσης από το ΕΓΚΕ με θέμα την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Όμως θα μου πείτε καλά όλα αυτά. Αλλά τι γίνεται με την εναρμόνιση, με τη συμφιλίωση επαγγελματική και οικογενειακής ζωής των γυναικών. Επειδή πιστεύω ακράδαντα, επειδή πιστεύουμε ακράδαντα στη γραμματεία ισότητα, ότι η ισότιμη γυναική συμμετοχή στην ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι δυνατή χωρίς τη συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, με μεγάλη μας χαρά στηρίζουμε τη διοργάνωση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στις 29 Απριλίου στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση υλοποιείται από τη Συνομοσπονδία Οργανώσεων για την Οικογένεια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείπει από τον διάλογό μας από την ατζέντα, ένα πάρα πολύ, μας ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που ταλαιπωρεί ακόμη και την Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο Αναφέρομαι στο θέμα της βίας κατά των γυναικών. Γι' αυτό το λόγο λάβαμε στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας ειδική μέρημνα για πολιτικές που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών και ιδιαίτερα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που τελικά εμφανίζει έξαρση, ιδιαίτερα στη φάση της οικονομικής κρίσης και μας απασχολεί έντονα σε εθνικό επίπεδο. αναγνωρίζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση όμως του προβλήματος αυτού η ελληνική προεδρία και ο οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης το γνωστό φρα διοργανώνουμε ειδικό θεματικό συνέδριο υψηλού επίπεδου ε, στις 5, Φεβρουαρίου, συγγνώμη, στις 5 Μαρτίου συγγνώμη, στις Βρυξέλλες όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης που εκπώνησε ο ΦΡΑ, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βία κατά των Γυναικών. Θα ήθελα εδώ, θα ήταν παρέλειψή μου, αν δεν τόνιζω ότι στο συγκεκριμένο τομέα υπάρχει ήδη μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Ιταλική κυβέρνηση. Μια συνεργασία που θα συνεχιστεί όταν η Ιταλία λάβει από τη χώρα μας, από την Ελλάδα, τη σκητάλη της Προεδρίας, διασφαλίζοντας τη συνεπή συνέχιση των πολιτικών για την πρόληψη και την εξάλληψη της βίας. Δεν νοείται όμως όπως εύκολα θα μπορούσε κάποιος να πει, θα συμφωνούσα μαζί του. Πρωτοβουλία για την ισότητα των φύλων χωρίς νομοθετικό έργο. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων χωρίς να ενισχυθούμε από ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό, στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, προωθούμε την ένταξη θεμάτων ισότητας των φύλων στα κατά περίπτωση αρμόδια Συμβούλια Υπουργών. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει αφορά την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα οικονομικά κέντρα αποφάσεων. Στη συνεδριά του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, το γνωστό ΕΠΣΚΟ, θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί η έκθεση πρόοδου σχετικά με την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Στην Ελλάδα, η Γενική Γραμματεία ισότητα των Φύλων έχει ταχθεί με σαφή τρόπο υπέρ κάθε μέτρου που προωθεί την ουσιαστική ισότητα των φύλων μέσω της ανταλλαγής νοοτροπίας, πρακτικών και της νομοθεσίας βέβαια εφόσον απαιτείται. Με δεδομένο όμως ότι αποτελεί, πρόκειται για ένα θέμα με διαθεματικό χαρακτήρα, στην Ελλάδα αναλάβαμε πρωτοβουλία για τη βέλτιστη διαχείρισή του με τη συμμετοχή συναρμόδιων Υπουργείων και υλικών Φορέων Επίση, στο πλαίσιο εργασιών του ΕΠΣΚΟ, τον Ιούνιο, θα παρουσιαστεί το σχέδιο συμπερασμάτων που εκπονείται από την Ελληνική Προεδρία με θέμα και γυναίκε. Το σχέδιο συμπερασμάτων θα βασίζεται στα αποτελέσματα τη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΓΚΕ. Αναμένεται η υιοθέτηση από το Συμβούλιο του σχετικού σχεδίου συμπερασμάτων. Τέλο, στο επίπεδο του νομοθετικού πλαισίου, του νομοθετικού έργου και σχετικά με το ζήτημα τη βία κατά των γυναικών, αναμένεται η υιοθέτηση των συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την προσπάθεια αυτή της διάχυσης της αρχής της ισότητας των φίλων σε όλη την κοινωνία δεν μπορεί να απουσιάζει η νέα γενιά. Δεν μπορεί να απουσιάζει η νέα γενιά των κρατών μελών, δεν μπορεί να απουσιάζει η νέα γενιά της Ευρώπης. Δεν μπορούν να απουσιάζουν οι νέες και οι νέοι Ευρωπαίοι. Έτσι, γενική Γενικοί της Ισότητας των Φύλων συμμετέχουμε μαζί με το ΕΓΕ στην Πανευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία, το Youth Event, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 13 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Επιδιώκουμε μέσω του τρόπου αυτού να μπορέσουμε να αγγίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους με τα μηνύματά μας. Να αναδείξουμε τις παγίδες του σεξισμού που κρύβει το διαδίκτυο τα αρνητικά έμφυλα στερεότυπα που αναπαράγουμε μέσα από το λόγο και την εικόνα. Να πάρουμε με το μέρος μας τους νέους άνδρες στον αγώνα αυτό για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών όσο υπάρχει ακόμα καιρός. Πριν το παιχνίδι της αντιπαλότητας των φίλων που ξεκινάει σχεδόν από το σχολικό προάβλιο παγιωθεί σε στάσεις και πράξει στην ενήλικη ζωή. Κάπου εδώ τελειώνουν οι δράσεις μας για την ελληνική προεδρία αλλά στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου γιατί θα ήταν μεγάλη παράληψη από την πλευρά μου να μην σταθώ στην πολύτιμη συμβολή των ευρωπαϊκών οργάνων σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση και υλοποίηση του προγράμματο τη ελληνική προεδρία στο τομέα τη ισότητα των φύλων. Για τον λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Μονάδα Ισότητα των Φύλων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γραμματεία του Συμβουλίου, το ΕΓΕ και το ΦΡΑ. Η συμβολή του, πιστέψτε με, ήταν ουσιαστική και καθοριστική για μα. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εταίρους μας στην Τριαδική Προεδρία που ολοκληρώνεται αυτό για το εξάμεινο, τους ομολόγους μου από την Ιρλανδία και τη Λιθουανία για τη συνεργασία και τη σύμπνοια που επέδειξαν. Τελειώνοντας, θα ήθελα ακόμα δύο-τρία λεπτά από το χρόνο σας. Three or more <laughs> και θα ήθελα να σταθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Μιλώντας ως ένας πολίτης της Ευρώπης επίσης, φανατικά φιλοευρωπαϊστής. Τελευταία πενταετία, κυρίες και κύριοι, της οικονομικής κρίσης ήταν σκληρή για την Ευρώπη και ακόμα πιο σκληρή για την πατρίδα μου. Ήταν ένα τεστ αντοχής που επιχειρήσαμε να, επιχειρήσαμε να περάσουμε χωρίς μεγάλα ρίσκα. Με συντηρητικές αποφάσεις, με επιφυλακτικότητα και χωρίς τελικά να πείσουμε κανέναν και κυρίως τους εαυτούς μας ότι η Ευρώπη έχει την πρόθεση να μείνει ενωμένη διαχρονικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε μου να πω, ότι εμφανίζεται σήμερα πολυδιασπασμένη και διχασμένη όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία της. Έχουν έρθει στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα που δημιούργησαν οι αποφάσεις που δεν πήραμε τελικά. Λείπει μια ισχυρή, ακλόνητη βάση για μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αντίθετα, κυριαρχεί ανεξέλεγκτη ιδεολογία του χρήματος, ένας στιγνός και κοινικός χρηματοοικονομικός ανταγωνισμός η ευρώπη δυστυχώς αδυνατεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ρυθμιστή να εξομαλύνει τις εντάσεις όπως έκανε παλιότερα. τίθεται τελικά σε αμφισβήτηση το πνεύμα στο οποίο βασίστηκε η ίδια η ευρωπαϊκή ιδέα. η απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων αγαθών υπηρεσιών και κεφαλαίων για κάποιους σήμερα θεωρείται απειλή. η αδράνεια κινδυνεύει να επιτρέψει στην ευρωπαϊκή ένωση να υποβαθμιστεί σε ένα χώρο ελεύθερων συναλλαγών υπαγκούοντας τελικά σε εθνοκεντρικές πολιτικές. Πού βρίσκεται άραγε η αντίληψη του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντο, όταν κάποιοι νιώθουν, κυρίε και κύριοι, φιλάνθρωποι και κάποιοι άλλοι αισθάνονται ότι ελεούνται. Ο πολίτη σήμερα, ο Ευρωπαίο πολίτη, νιώθει εγκατάλειψη, απογοήτευση για μια Ευρώπη που δεν καταφέρνει να λύσει τα προβλήματα και να προσφέρει δουλειέ και σταθερότητα. Δεν καταφέρνει να αποτελέσει μια ισχυρή ελπίδα απέναντι στι προκλήσει τη παγκοσμιοποίηση. Όμω, κυρίε και κύριοι, δεν είναι αυτό που οραματίστηκαν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για το οποίο μάθαμε στα φοιτητικά μας χρόνια. Αυτό για το οποίο αγωνιστήκαμε στα νεανικά μας χρόνια και φτάσαμε ως, σήμερα. Εκείνο των ιδρυτών των θεμελιωτών της ιδέας Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένα όραμα ειρήνης, σταθερότητας, ευημερίας και δημοκρατικών αξιών. Βασιζόταν στην πολιτική ένωση και εκφραζόταν με τους όρους ενός ιδεαλισμού που μπορούσε να συνεγείρει τους λαούς για θυμηθείτε την επιθυμία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, μόλις έπεσε το τείχος, να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμηθείτε τη μεγάλη διεύρυνση του 2003 που έγινε κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Για μια πραγματική αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης μιλούσε ο Σουμάν στην ιστορική διακήρυξη στις 9 Μαρτίου του 1950 την οποία γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Μια αλληλεγγύη που θα αναπτυσσόταν μέσα από απτά επιτεύγματα της Ευρώπης. Ο Αντενάουερ, απ' την άλλη, οραματιζόταν μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Ο Ντεκάσπερι, ο Ντεκάσπερι συγγνώμη, ήδη από το 1951 είχε δει το κίνδυνο. Λέει σε κάποια του ομιλία. Αν περιοριστούμε στη δημιουργία κοινών διοικήσεων χωρί μια ανώτερη κεντρική αρχή που θα συγκεντρώνει, θα διαμορφώνει και θα προάγει σε ένα ανώτερο επίπεδο τι εθνικέ επιδιώξει, υπάρχει κίνδυνο τα ευρωπαϊκά όργανα να μην έχουν πλέον καμία ουσιαστική αξία ή όραμα σε σύγκριση με τον δυναμισμό των διαφόρων κρατών. Θα μπορούσαν ακόμη και συνεχίζει να φτάσουν στο σημείο να θεωρούνται ως περιττοί και δεσμευτικοί θεσμοί όπως συνέβαινε και το τονίζει αυτό κατά την περίοδο της παρακμής της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι 60 χρόνια μετά τα λόγια αυτά ακούγονται προφητικά όταν η Ευρώπη φαίνεται προς τους πολίτες να έχει χάσει τον δρόμο της όταν κινδυνεύει να καταλήξει κάτι λιγότερο από το άθροισμα των μερών της να μετατραπεί σε ένα ενδιαφέρον αλλά αποτυχημένο πείραμα αν μπορούσα να το πω όπως το λέγαμε στα φοιτητικά μας χρόνια ενοποίησης της γυραιάς υπήρου. Γιατί τελικά η Ευρώπη, κυρίε και κύριοι, μπορεί να είναι ισχυρή μόνο μέσα από την ενότητά τη. Η Ευρώπη μπορεί να υπάρχει μόνο μέσα από την ενότητα των κρατών μελών της. Για τον λόγο αυτό, στι εκλογέ του Μαΐου δεν θα κρυθεί μόνο η δύναμη και η δημοφιλία του κάθε κόμματο στι χώρε μέλη. Θα κρυθεί το ίδιο το μέλλον τη Ευρώπη. Άραγε, ο πολίτη που θα προσέλθει στι Ευρω... κάλπε των ευρωεκλογών έχει μπροστά του σαφεί και ορατέ επιλογέ για το μέλλον τη Ευρώπη ή ακόμη και για το παρόν τη. Πόσο ξεκάθαρη αισθάνεται τελικά την ευρωπαϊκή του ταυτότητα για την οποία κάποτε μιλούσαμε. Υπάρχει κάτι που συνεχίζει πραγματικά να μας ενώνει, παρά τις αντιπαραθέσεις, παρά τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές μας. Με συγχωρείτε, αλλά έχω την εντύπωση, έχω την αίσθηση ότι τα ερωτήματα αυτά ακόμη και σήμερα δεν έχουν απαντηθεί. Γιατί αν είχαν απαντηθεί θα είχαμε τελικά αποφασίσει αντίστοιχα τι δεν είναι Ευρώπη. Συνά στρέφω το βλέμμα μου γύρω και διερωτώ με αν μοιράζομαι με το διπλανό μου ή τη διπλανή μου την ίδια αντίληψη, τις ίδιες προσδοκίες, τις ίδιες αξίες για την κοινή αυτή περίφημη Ευρώπη. Αν μοιραζόμαστε τελικά μια κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση. Αν πράγματι μας συνδέουν κοινέ ιστορικές αναφορές, για παράδειγμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στο μοντέλο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στη ρωμαϊκή λατινική χριστιανοσύνη, στο ορθόδοξο Βυζάντιο, στη νομική κληρονομιά του Καρλομάγνου, στους πρώτους κοινούς οικονομικούς χώρους του Μεσαίωνα Άραγε αισθανόμαστε όλοι δικό μας το διαφωτισμό και το κοσμικό απελευθερωτικό του πνεύμα, τη Γαλλική Επανάσταση, τον Ευρωπαϊκό Ανθρωπισμό, τη πίστη στη γνώση και στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Μια νέα Ευρώπη, μια ήπειρος των πολιτισμών και των πολιτών μπορεί και πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Το όραμα για μια νέα Ευρώπη βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής χρειάζεται πολιτικές συνειδητής αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη, σε βορρά και νότο, κέντρο και περιφέρεια ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές αλλά και ανάμεσα στα δύο φύλλα για να γυρίσουμε στα δικά μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε στη δημιουργία μιας κοινή Ευρώπης. Η κρίση έχει ήδη προσφέρει πάρα πολλά αντιευρωπαϊκά επιχειρήματα σε πολλές και ποικίλε φυγόκεντρες δυνάμεις. Δυστυχώς ο ευρωσκεπτικισμός κερδίζει έδαφος. Μέσα σε ένα περιβάλλον αμφισβήτηση και κριτικής αναδεικνύονται και κάποιες άλλες φωνές, ακραίε κερδίζουν έδαφο μορφώματα και δυναμικέ μια φοβική εσωστρέφεια και μυσαλλοδοξία. Η νεκρανάσταση του φασισμού και του ναζισμού πυροδοτεί νέε κοινωνικέ εντάσει. Παρασύρει τμήματα τη κοινωνία που σήμερα βιώνουν την απογοήτευση και την απόγνωση. Κινδυνεύουμε τελικά να γίνουμε μάρτυρες μιας σταδιακής κατάλυσης όλων των ευρωπαϊκών μας αξιών. Στη προσπάθεια αυτή για την ενωμένη ήπειρό μας, για τη μια ήπειρο των πολιτών, η ευρώπη χρειάζεται το 100% του δυναμικού της. οι δημιουργικές δυνάμεις της γυναίκας μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην έξοδό μας από την κρίση από μια κρίση που επιτρέψτε μου να πιστεύω και να πω και να στηρίζω ότι δεν είναι μόνο οικονομική αλλά είναι παράλληλα μια κρίση αξιών και μια κρίση αρχών. είναι κρίση κοινωνική και πολιτισμική είναι κρίση ηθική εν τέλει. στην ελλάδα για το λόγο αυτό υλοποιούμε μια μεγάλη εκστρατεία για την ισόρροπη συμμετοχή υποψηφίων και των δύο φύλων στα κέντρα αποφάσεων τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιδιώκουμε θερμότερη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στι ερχόμενε ευρωεκλογέ. Του ζητούμε να επιλέξουν περισσότερε γυναίκε σε μια περίοδο κρίσιμη για τη χώρα μα, αλλά ταυτόχρονα κρίσιμη και για τη τύχη ολόκληρη τη Ευρώπη. Α ελπίσουμε και εύχομαι ταυτόχρονα το 2014, κυρίε και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγγνώμη κύριε Πρόεδρε γι' αυτό, να αποκτήσει ακόμα περισσότερες γυναίκες. Γιατί έχει αποδείξει ότι είναι εκείνο ο θεσμός που λειτουργεί ως ο θεματοφύλακα σημαντικών αξιών του πολιτισμού μας. Αξιών πάνω στις οποίες μπορεί να οικοδομηθεί μια Ευρώπη των πολιτών. Φίλε και φίλοι, θα ήθελα να τελειώσω με, τούτη, με τούτο. Γιατί κάποιε φορέ κάποιοι μου λένε ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον τη Ευρώπη. Ενώ κάποιοι πιστεύουν ότι η Ευρώπη διανύει τι τελευταίε τη μέρε. Το να ελπίζει σε δύσκολου καιρούς δεν είναι ανόητα ρομαντικό. Είναι βασισμένο στο γεγονό ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι μόνο μια ιστορία σκληρότητα. Είναι ταυτόχρονα μια ιστορία συμπόνια, θυσία, θάρρου, καλοσύνη και αλληλεγγύη. Και με αυτό, με αυτή την ελπίδα και το τρόπο και για ποιο λόγο στηρίζομαι σε αυτή την ελπίδα θα ήθελα να κλείσω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας σήμερα εδώ, για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για τα εισαγωγικά σας λόγια. Ξέρω Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις σε εσά, αλλά πριν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια σημαντικά σημεία που αναφέρατε. Η στρατηγική 2020 και ο στόχος της απασχόλησης το 25% είναι κάτι που έχει συζητήσει πολλά και σε αυτή η Επιτροπή και έχουμε πετύχει το στόχο αυτό σε ό,τι αφορά τους άνδρες, αλλά δεν έχουμε πετύχει το στόχο αυτό σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες συνεχίζουν να είναι οικονομικά εξαρτημένες και πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά θα λειτουργήσουν στο μέλλον και να εξετάσουμε και αυτή την ε, πτυχή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τις υπηρεσίες πρόνοιας, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Και αν δεν ε, είσαι οικονομικά ανεξάρτητος, ε, δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις για τη ζωή σου. Επομένως, αυτές είναι πολύ σημαντικές πτυχές, όπως είπατε και εσείς. Κάτι άλλο που αναφέρατε που είναι ουσιώδες είναι ότι ποτέ δεν ε, βλέπουμε την ποιότητα ως κόστος. Αν θέλουμε να πετύχουμε την ε, ποιότητα θα πρέπει να σκεφτούμε την ανάπτυξη της κοινωνίας, θα πρέπει να κινήσουμε την ε, κοινωνία προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να σκεφτούμε την ισότητα όχι ως κόστος αλλά αν η κοινωνία αναπτύσσεται και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε αυτό είναι όφελος. Ε, τώρα, αναφερθήκατε σε δύο διασκέψεις. Ε, μία θα γίνει τον Απρίλιο και έχουμε και την διάσκεψη της 5ης Μαρτίου. Εκεί θα παρουσιαστεί μία πολύ μεγάλη μελέτη και τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής και θα συζητηθούν και σημαντικά θέματα που έχουμε συζητήσει και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, έτσι λοιπόν, κατόπιν αυτών των σύντομων σχολείων από πλευρά μου θα ήθελα να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ε, συναδέλφους, η κυρία Μπάστος καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Ελληνική Προεδρία και να ευχηθώ καλή επιτυχία για το επόμενο εξάμεινο. Επίσης ευχαριστώ την κυρία Γενική Γραμματέα, την κυρία Κόλια, για την παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Προεδρίας για την ισότητα των φύλων. Αναφερθήκατε σε διάφορα σημεία που μας απασχολούν και μας αυτή την Επιτροπή. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην ε, βάση της επίτευξης, της προόδου που θεωρούμε εμείς ότι είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να έχει ίσες ευκαιρίες και η γυναίκα στην κοινωνία, σε όλα τα επίπεδα, θα ήθελα εγώ να μάθω το εξής. σε σχέση με την ε, επιρροή που μπορεί να ασκήσει η ελληνική προεδρία στο συντονισμό πολιτικών σε επίπεδο ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών, αν η ψηφιακή οικονομία, στην οποία αναφερθήκατε ως ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της ισότητας, ε, μήπως ε, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό το μεγάλο στόχο της συμφιλίωσης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να τονίσω είναι στο πλαίσιο της κρίσης που βιώνουμε σε ορισμένα κράτη-μέλη και κυρίως στην Νότια Ευρώπη, αναφέρομαι στην οικονομική, χρηματοπιστωτική κρίση, στο θέμα της απασχόλησης. Δεν ε, υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες ε, σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να μου πείτε αν η ελληνική προεδρία είναι ευαισθητοποιημένη απέναντι σε κάποια είδη βίας που αρχίζουν να αναδύονται και ιδίω στο διαδίκτυο και κυρίως σε σχέση με τις διάφορες ηλικιακέ ομάδες και επίσης ε, τι συμβαίνει στα πλαίσια των οικογενειών που βιώνουν την οικονομική κρίση και θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα στο Κοινοβούλιο, το οποίο έχει να κάνει με την ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως ξέρετε, το Κοινοβούλιο με μεγάλη σαφήνεια τοποθετήθηκε στην ε, ψηφοφορία του ψηφίσματος στην Ολομέλεια και δεσμεύτηκε ισχυρά υπέρ αυτής της εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλών επιχειρήσεων. Εμεί θεωρούμε ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ρεαλιστική και ισορροπημένη και ότι το Συμβούλιο επομένως έχει μία καλή βάση για να συνεχίσει αυτή την εργασία και για να ολοκληρωθεί ο φάκελος αυτός κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε αν η ελληνική προεδρία θα πολεμήσει για το φάκελο αυτό, θα προσπαθήσει να επηρεάσει τους συναδέλφους σας, θα προσπαθήσει να επηρεάσει τους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο, έτσι ώστε να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Και η κυρία Κράτσα που δεν μπορεί να παρευρεθεί αυτή τη στιγμή εδώ, θέτει αυτή την πρόταση. Ότι η ιδέα που έχουμε εμείς είναι ότι θα έχουμε υποστήριξη και ότι θα ήθελα να ξεκαθαρίσω αυτό και ότι οι επόμενες ευρωεκλογέ θα είναι ένα σημαντικό βήμα, ένα σημαντικό μήνυμα για τους πολίτες μας, έτσι ώστε να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράγματι έχει αναλάβει δεσμεύσεις, έχει δεσμευτεί να εμβαθύνει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Αυτές τις ερωτήσεις θέλω να θέσω εγώ. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκουρμά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κόλια για τις βαθιές πεπιθήσεις σας για το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Πάντα είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να καλωσορίζουμε άτομα τα οποία είναι στρατευμένα στον αγώνα αυτό τη ισότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης που μπορούμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την ελληνική προεδρία, γιατί με τον τρόπο αυτό κλείνει ο κοινοβουλευτικό ε, κύκλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρουμε ότι θα τελειώσει η θητεία του Κοινοβουλίου ουσιαστικά στις 18 Απριλίου, αλλά πρέπει να συνεχίσει το έργο αυτό γιατί το πρόγραμμα της, της Ελληνικής Προεδρίας και της φιλοδοξίας σας σε ό,τι αφορά την ισότητα των φίλων Είναι πάντα πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η ισότητα αυτή ως όχι μόνο θεμελιώδης αξία, αλλά ως κινητήρια δύναμη για να μπορέσει να υπάρξει απόλυτη ισότητα στον κοινωνικό χώρο <clears throat> και η Ισπανική Προεδρία έχει τονίσει πάρα πολύ το στόχο αυτό. Χαίρομαι επίσης επειδή αναφερθήκατε στην ε, ανάγκη να εστιάσουμε περισσότερο στο ρόλο των γυναικών στην οικονομία και επίσης χαίρομαι με την συνεργασία σας με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Νομίζω ότι ο ρόλος του είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικός εν ώψη και της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής μας για, την, για τα θέματα αυτά. Θυμάστε ότι στη στρατηγική της Λισαβόνας είχαμε συγκεκριμένους στόχους και για τους άντρες και για τις γυναίκες ενώ υπάρχει ο στόχος της απασχόλησης, του ποσοστού απασχόλησης 75% στη στρατηγική 2020, ενώ ξέρουμε ότι οι γυναίκες υπολείπονται, βρίσκονται στο 60-62% ενώ οι άντρες έχουν πετύχει βασικά αυτό το στόχο. Έχουμε πολλά να κάνουμε λοιπόν για να επιτύχουμε την ισότητα στο χώρο αυτό και μέσα σε αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να τα πράξουμε αυτά αν θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτή την δέσμευση που αναλάβαμε το 2010. Χρειαζόμαστε πιο επακριβείς επίσης δείκτες σε σχέση με την επιτυχία του λεγόμενου gender mainstreaming, της εισαγωγής της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Αυτή η πολιτική του mainstreaming μπορεί να οδηγήσει σε προσθέμενη αξία σε όλους τους τομείς πολιτικής. Αναφερθήκατε, ε, αναφερθήκαμε και στην Επιτροπή μας, συγγνώμη, στο θέμα του Ινστιτούτου Ισότητος για τα θέματα αυτά. Επίσης, η συνδιάσκεψη στην οποία αναφερθήκατε θα πρέπει να ακολουθηθεί από συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Αυτό είναι απαραίτητο. Και επίσης χαίρομαι για τα συμπεράσματα που αναφέρατε για την ανάγκη να υπάρξει συνέχεια στα συμπεράσματα του Συμβουλίου έψω του και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ουσιαστικές ενέργειες και όχι απλώς δηλώσεις. Και τέλος, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ακολουθώ αυτά που είπε η κυρία Μπάστος, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για την οδηγία περί ίσης διαχείρισης και το να υπάρχει ισότητα βάσει ποσοστώσεων στις διοικητικές θέσεις που δεν είναι εκτελεστικού χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό και για τις δύο πλευρές γιατί όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι όταν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες οι οποίες ε, εμπλέκονται σε αυτές τις θέσεις έχουμε όλοι να κερδίσουμε κάτι. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα της ανεργίας σε χώρες όπως η Ελλάδα που ξεπερνάει το 60%. Όταν οι νέοι δεν περιμένουν να έχουν ένα μέλλον σε αυτή την Ευρώπη, φυσικά θα στραφούν εναντίον της. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια σαφή δέσμευση για τα θέματα αυτά. Και ακούγοντα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο για να επιβιώσουμε ως Ευρώπη. Εσείς τονίσατε την προσωπική σας δέσμευση, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κρατήσουμε ζωντανή την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Κονέλσεν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κόλια. Την... Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Επανέρχομαι σε αυτά που ανέφερε η κυρία Μπάστος για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και την αντίστοιχη ε, οδηγία. Το γεγονός ότι διορίστηκε μία Γερμανίδα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας, αυτό είναι μία σημαντική πρόοδος και υπήρχε και μία γαλλική πρόταση να συμφωνήσουν για να υπάρξει μια κοινή εντολή διαπραγμάτευσης για την εντολή αυτή. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι θα κάνει η ελληνική προεδρία για να, προ... για να καταφέρει να μεταπίσει τη Γερμανία και να τη φέρει από αυτούς που εμποδίζουν την υλοποίηση αυτής της οδηγίας σε αυτούς που θέλουν να την εγκρίνει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει από τη δική σας πλευρά μια αναλλακτική πρόταση που να βασίζεται στην γαλλική θέση, που να μπορέσει να πει στη Γερμανία και φυσικά και μια άλλη χώρα. Επίσης η οδηγία για την μητρική άδεια η Ιρλανδική Προεδρία προσπάθησε να επιτύχει κάποια πρόοδο στα θέματα αυτά και φάνηκε να υπάρχει κάποια πρόοδος και από την πλευρά του Συμβουλίου και από τη δική μας πλευρά. Εμείς βέβαια από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήμασταν πάντα έτοιμοι να προβούμε σε συμβαστικές λύσεις και αυτός είναι ο στόχος των τριλόγων. Αλλά κάπου πρέπει να βρεθεί αυτή η ενδιάμεση συμβαστική λύση η Ελλαδική Προεδρία ακολούθησε μια κάπως παράξενη διαδικασία για το θέμα αυτό και τελικά δεν επέτυχε γιατί ήταν πραγματικά παράδοξη διαδικαστικά η διαδικασία. Θα δώσει λοιπόν μια νέα όθηση η Ελληνική Προεδρία. Βρισκόμαστε βέβαια στην απαρχή της Προεδρίας, αλλά ίσως με τις δικές σας προσπάθειες θα μπορέσει να επιτευχθεί κάτι. Και επίσης η η οδηγία εναντίον των διακρίσεων η ελληνική προεδρία θα διερευνήσει αν με τη νέα κυβέρνηση στη Γερμανία δεν θα υπάρχει πια στάση εμπλοκής από την πλευρά της Γερμανίας, αλλά υπάρχει δυνατότητα πρόεδρου. πρόοδου. Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει μια αξιολόγηση του έργου της Τρόικα, αλλά αυτό δεν αντιμετωπίζεται υπό την οπτική γωνία της ισότητας των φύλων, όπου εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σημαντική επίπτωση αυτών των προγραμμάτων για την ένδια, για τις ε, ε, περικοπές στην υγεία, στις δημόσιες δαπάνες. Νομίζω ότι η ελληνική προεδρία είναι σε πολύ καλή θέση να εξασφαλίσει ότι περιλαμβάνεται σε αυτή την αξιολόγηση και το θέμα της ισότητας των φύλων. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη θα πρέπει να σας ζητήσω γιατί καθυστέρησα λιγάκι. Έχω μόνο τρεις συναντήσεις επιτροπών που συμβαίνουν παραλίλω, που λαμβάνουν χώρα παραλίλως. Δεν μπορώ να είμαι πανταχού παρούσα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα σε σχέση με αυτά που αναφέρατε. Από ό,τι γνωρίζω, επειδή η δική μας πρώτη προτεραιότητα είναι η νομοθεσία και ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη αντίθεση στο Συμβούλιο, όχι μόνο μια μειοψηφία ανάσχεση, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη ομάδα κρατών που δεν θέλουν να υπάρξει νομοθεσία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση. Πώς θα θέλατε να αντιμετωπίσετε με το ζήτημα αυτό ποια είναι η προοπτική που βλέπετε να ανοίγεται μπροστά σας, θεωρείτε ότι θα μπορέσει το θέμα αυτό να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας ή όχι. Ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Γνωρίζουμε ότι εφέτος είναι το έτος το οποίο είναι αφιερωμένο στην συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Από ό,τι είπατε, ήδη έχετε προγραμματίσει μια συνδιάσκεψη για το θέμα αυτό. Πέραν αυτού θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποιες ιδέες που θα ε, θέσετε για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελόνης σε σχέση με τις προϋποθέσεις για την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. και φυσικά είναι βραχία η ελληνική προεδρία. Αναφέρατε ότι θα έχετε μια εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο. Για να προωθήσετε περισσότερες γυναίκες στα Ευρωψηφοδέλτια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναρωτιέμαι αν έχετε κατά νου κάτι αντίστοιχο ως Προεδρία του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. κυρία Μορβάη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας πω ότι είμαι αρκετά απογοητευμένη. Είστε μια γυναίκα από την Ελλάδα και εγώ νόμιζα ότι θα αποτελούσατε μία φωνή για όλες τις καταπιεσμένες γυναίκες ε, που υποφέρουν τα μάλα ε, λόγω αυτής της ε, πολύ άδικης οικονομίας και όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Τρόικα. Όμως οι αδελφές σας στην πατρίδα σας υποφέρουν πάρα πολύ και φυσικά και δικές μου αδελφές στη δική μου πατρίδα, στην Ουγγαρία. Εγώ θεωρούσα ότι θα ήσασταν ε, μία φωνή για τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή για χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, οι πρώην κομμουνιστικές χώρες όπου οι γυναίκες βρίσκονται δύο φορές σε πιο δινή θέση και επειδή είναι γυναίκες αλλά και επειδή προέρχονται από μειονεκτικές και σχεδόν ε, ε, χώρες απικίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ άκουσα εσάς να ε, παρουσιάζετε κάποια εγκόμια εδώ στην Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ανήκω στην ευρύτερη ομάδα των ευρωσκεπτικιστών, αλλά προσπαθώ να είμαι ανοιχτή απέναντι στα επιχείρηματά σας. Όμως μπορώ να πω ότι δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Προέρχεστε από μια χώρα όπου έχουμε 60% ανεργία στους νέους και πάρα πολλές γυναίκες φανταζόμαι υποφέρουν από την ανεργία και είναι και μητέρες. και οι οποίες ε, φυσικά επιφέρουν γιατί εγκαταλείπουν τη χώρα τα παιδιά τους και μπορούν τελικά να επικοινωνήσουν μαζί τους μόνο με το Skype. Θα σας παρακαλούσα να μας πείτε Δύο λόγια παραπάνω για τα αποτελέσματα των οικονομικών περιορισμών στις γυναίκες της χώρας σας και να μας πείτε δύο λόγια για το τι θέλετε να κάνετε ως ελληνική προεδρία προκειμένου να αντιμετωπίσετε τα τραγικά προβλήματα των γυναικών που βρίσκονται σε ανέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανεργία των γυναικών ιδίως και τα αποτελέσματα της κρίσης. Και γιατί νομίζετε ότι αν ενδυναμωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτική ένωση αυτό θα συμβάλλει και στην ισότητα των γυναικών. Εμείς το αντίθετο βλέπουμε. Δηλαδή πώς συγκρίνεται την κατάσταση μιας γυναίκας στην Νορβηγία με μια γυναίκα στην Ελλάδα. Η Νορβηγία δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ε, δεν βλέπω να υποφέρουν οι γυναίκε εκεί επειδή δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ όλα αυτά συνάδουν λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ισότητα των δύο φύλων. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε κάτι για την ανέχεια που βιώνουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κολλή να απαντήσει στα σχόλια και τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Αγαπητό αξιότιμο μιλούσε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς θεωρώ ως απλός πολίτης, Ευρωπαίος πολίτης, με εθνική μένει ταυτότητα, ελληνική ταυτότητα, αλλά νιώθω τον εαυτό μου Ευρωπαίο πολίτη, ότι όσοι είμαστε εδώ μέσα ή ασχολούμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δουλεύουμε πάντοτε προ τη θετική κατεύθυνση και για το καλό των λαών μα, Άλλωστε, όπω ανέφερα και πριν, η ιστορία μα έδειξε ότι μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου του 1989, όλε οι χώρε οι οποίε άνοικαν στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ έσπευσαν να γίνουν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάτι λέει. Αν σήμερα έχουν γίνει κάποια λάθη, τα οποία κανεί δεν μπορεί να αρνηθεί και στην περίπτωση τη χώρα μα, σίγουρα υπάρχουν λάθη τα οποία έχουμε κάνει εμεί. Υπάρχουν όμως λάθη, όπως όλοι μας παραδεχόμαστε, και στο κατασκευαστικό αυτό οικοδόμημα του ευρώ. Σίγουρα υπάρχουν λάθη, όπως σας είπα, και στις πολιτικές που πλέον μπορεί να έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει δώσει μεγαλύτερη σημασία στην οικονομία παρά στους ανθρώπους και στην πολιτική, η οποία έχει δώσει μεγαλύτερη σημασία σε μια οικονομία άειλη, σε μια οικονομία χρηματοοικονομική, στο ε, χρηματοοικονομικό κομμάτι, παρά στην πραγματική παραγωγή, την οποία παραγωγή έχει στείλει σε άλλε χώρε. Άρα το να εκ των προτέρων να στεκόμαστε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην φροντίζουμε να διορθώσουμε τα κακό σημερινά κείμενα, επιτρέψτε μου να πω θα διαφωνήσω μαζί σας. Απλά πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό αναφέρθηκα στους ιδρυτές, να γυρίσει πάλι πίσω στις αξίες με τις οποίες οικοδομήθηκε και χώρε σαν τη δική μου, μικρή χώρα, χώρε σαν τη δική σα, θελήσαμε να γίνουμε μέλη. Η χώρα μου, δεν σα κρύβω, κέρδισε και ευεργετήθηκε σε πολλά σημεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις γυναίκες, τόσο οικονομικά όσο και νομοθετικά. Πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν θα έχει προχωρήσει αυτό, μπορεί και να έχει προχωρήσει. Άποψή μου είναι πως όχι. Το οικογενειακό δίκαιο που έχουμε σήμερα και δίνει μία ισότιμη θέση της γυναίκας στην ελληνική, οικονομία, στην ελληνική κοινωνία και της δίνει δικαιώματα προήλθε από τη συμμετοχή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, για μένα η θέση μου και η θέση τη ελληνική προεδρία θα είναι να παλέψουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε, αφήνοντα πίσω τα άσχημα σημεία, τα σημεία που όλου μα στενοχωρούν και όλου μα έχουν φέρει σε δύσκολη θέση και ακόμα περισσότερο τη χώρα μου. Ε, να προχωρήσω τώρα, αφού ξεκίνησα από το τέλος, θα συνεχίσω από το τέλος. Ε, σχετικά με την οριζόντια οδηγία εναντίον των διακρίσεων. Θέλω να σας πω ότι η Ελληνική Προεδρία, τόσο η Γραμματεία Ισότητας αλλά και το Υπουργείο Εργασίας, που ε, αν συμμετάσχετε αύριο νομίζω παρουσιάζει το πρόγραμμα της Προεδρίας ο καθήλυνα αρμόδιος Υπουργός, θα ασχοληθούμε κατά των διακρίσεων. Κατά διακρίσεων Αυτό Θα και θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ε, θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με το άρθρο 2 που αφορά την έννοια της διάκρισης. Ε, έννοια της Το θέμα αυτό θα αρχίσει, ε, όπως γνωρίζουμε, θα εξεταστεί πρώτα από την ομάδα κοινωνικών θεμάτων και μετά θα πάρει την σειρά που πρέπει να πάρει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με, το, με, τις, γονικές άδειες, θέλω να σας πω ότι καταρχάς είμαστε απόλυτοι σύμφωνοι και ο ιδιαίτερος γυναίκα δεν θα μπορούσα να διαφωνούσα ε, σε κάτι τέτοιο. Για τη χώρα μου ίσως τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα γιατί όπως γνωρίζετε δεσμευόμαστε από το πρόγραμμα της Τρόικας, το πρόγραμμα το οποίο ακολουθούμε. Ως Προεδρία όμως ε, θέλουμε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Ε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που διαφωνούν. Ε, εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανασύρουμε πάλι το θέμα από το ράφι, να προχωρήσουμε αλλά ίσως και η χρονική συγκυρία και εδώ είναι και ένας προβληματισμός δικός μας η χρονική συγκυρία καθότι η ελληνική προεδρία όπως και εσείς αναφέρατε είναι μικρής διάρκειας λόγω των ευρωεκλογών να μην είναι και καταλληλότερη και δεν θα θέλαμε ίσως να ξεκινήσουμε ένα θέμα μειώντας σίγουρο ότι θα έχει ε, θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση που όλοι επιθυμούμε. Ε, το αφήσω τελευταία για την κρίση. Επειδή ετέθη το θέμα της κρίσης, νομίζω ότι απάντησα στην αρχή και ε, νομίζω σας έχω καλύψει. Αυτή, αν θέλετε, είναι και η προσωπική μου άποψη, ότι η Ευρώπη πρέπει να ξεφύγει από αυτό το κομμάτι της άλλης οικονομίας, πρέπει να φέρει ξανά στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και την πολιτική και η οικονομία να είναι απλά εργαλείο για την ευτυχία και την ευημερία των λαών της Ευρώπης. Άλλωστε γι' αυτό φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι θα επαναλάβω για την ευημερία, την αλληλεγγύη και τη συναδέλφωση των λαών της. Σχετικά με τη συμφιλίωση επαγγελματική και οικογενειακής ζωής και τη σχέση με την ψηφιακή οικονομία. Ε, δεν χρειάζεται να, να, να το υποστηρίξω με κάποιο δυνατό επιχείρημα γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι οι γυναίκες εκείνες που έχουν παιδιά ή άλλες υποχρεώσεις και λόγω της κρίσης δυστυχώς εκτός από τα παιδιά τους φορτώνονται όπως ήδη σας ανέφερα και με άλλες υποχρεώσεις να προστατεύουν να φροντίζουν τους γονείς ή μεγαλύτερους ανθρώπους, σαφώς τις διευκολύνει να είναι ενεργές, να είναι δυναμικές στο οικονομικό και κοινωνικό κομμάτι, αν τους δίνεται η δυνατότητα να φτιάξουν μια επιχείρηση μέσα από το διαδίκτυο ή να κάνουν τη δουλειά τους μέσα από το διαδίκτυο. Γι' αυτό αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς στόχους που προωθούμε την ψηφιακή οικονομία στο κομμάτι τουλάχιστον κατά εμά του γυναικείου πληθυσμού. σχετικά με το θέμα της βίας. Όπως ήδη σας είπα, στις 5 Μαρτίου, σε συνεργασία με το ΦΡΑ, θα παρουσιάσουμε την έρευνα που έχει εκπονήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εδώ στις Βρυξέλλες. Ήδη πριν λίγο πήρα μια πρόσκληση για την ίδια ημέρα στις 7 το απόγευμα εδώ για να μιλήσουμε πάλι για το θέμα της βίας. Στην Ελλάδα να σας πω, το θέμα της βίας δεν είχε αναδειχθεί επαρκώς όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ένα από αυτά τα προβλήματα και νομίζω το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το σπρώχνουμε κάτω από το χαλί. Αυτό που θα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες τα ενίκου μη ενδύμου. Δυστυχώς τα ακολουθούμε σε αυτό το πρόβλημα. Ε, σκοπός μας είναι μετά την έρευνα και περνώντας τα συμπεράσματα και στο Συμβούλιο Υπουργών ε, να σχεδιάσουμε μία δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τόσο τις γυναίκες που, θύμα, που είναι θύματα βίας, αλλά και τους άνδρες. Όχι τους άνδρες απαραίτητα που είναι θύτες και προσπαθούν οι κύριοι πολλές φορές να ξεπεράσουν το πρόβλημα, αλλά και τους άνδρες, στο γενικό πληθυσμό των ανδρών, γιατί τουλάχιστον αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε στην Ελλάδα είναι σε κάθε πρωτοβουλία που παίρνουμε να έχουμε δίπλα μας και τον ανδρικό πληθυσμό, γιατί πιστεύουμε ότι ισότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γυναίκες και άνδρες ισότητα μπορεί να υπάρξει μόνο με τη συμμετοχή και την προσπάθεια και των δύο φίλων. Ε, θα ήθελα, αν είχατε λίγο χρόνο, να σας πω σε αυτά που κάνουμε τουλάχιστον στην Ελλάδα ότι έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο 40 συμβουλευτικών κέντρων για γυναίκες θύματα βίας και 21 φιλο... ε, ξενώνες φιλοξενίες για τις γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους. Ταυτόχρονα ε, έχουμε θέσει λειτουργία εδώ και δυόμιση περίπου χρόνια ε, μία τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας, 24 ώρες λειτουργίας. Ε, η, ε, γραμμή, η γραμμή έχει το νούμερο 15900 και είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια γραμμή hotline. όπου απευθύνονται οι γυναίκες για την πρώτη βοήθεια, την πρώτη στήριξη. Πληροφορίες δίνονται και στα αγγλικά. η γραμμή έχει δεχτεί μέχρι σήμερα, ίσως το νούμερο σας φανεί μικρό, περίπου 12.500 κλήσεις. Ε, αλλά θα ήθελα να κρατήσετε ότι είναι 12.500 κλήσεις σε μια χώρα, σε μια μικρή χώρα με πληθυσμό 10 εκατομμύρια πολίτες περίπου. Ε, πέραν αυτού του, αριθμού που σας ανέφερα, είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, ένας σκοτεινός αριθμός πίσω από τις κουρτίνες γυναικών που ακόμα δεν τολμά να καταγγείλει την βία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να φέρουμε αυτές τις γυναίκες στο φως, να τις βοηθήσουμε να έρθουν να καταγγείλουν την βία και να πάψουν να ντρέπονται ή να φοβούνται το κοινωνικό περίγυρο. Αυτό όμω το στερεότυπο, αυτή η να φοβουνται το κοινωνικο περιγυρο αυτο ομως νομίζω θα πρέπει να την δούμε όλοι μαζί, γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είμαι βέβαιη ότι αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να γυρίσω στο πολιτικό κομμάτι της ομιλίας μας, δεν εννοείται η Ευρώπη της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, η Ευρώπη του ρωμαϊκού δικαίου, η Ευρώπη του διαφωτισμού, το 2014 να μην μπορεί ακόμα να λύσει το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Ε, τι άλλο είχαμε, τι κρίση, ε, τα Ναι, δεν για να περάσουμε τώρα στο μεγάλο θέμα, το οποίο μάλλον ταλαιπωρεί όλους μας και ίσως επιτρέψτε μου να πω ανθρώπινα, εμένα ακόμα περισσότερο, γιατί μόλις ανέλαβα περίπου 7 μήνες έπρεπε να το αντιμετωπίσω αμέσως και εννοώ την πρόταση οδηγίας για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των, των εκτελεστικών οργάνων των εταιριών. Ε, όπως ήδη γνωρίζετε, η διαπραγμάτευση αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Θέλω καταρχά να σας πω, το έχω πει και στην κυρία Κράτσα, ε, το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός της χώρας και σκοπός της Προεδρίας, της Ελληνικής Προεδρίας, το θέμα αυτό θα ήταν να κλείσει, να κλείσει με επιτυχία. Ε, αλλά μελετώντας το συνεχώς, ε, πολύ φοβούμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση διότι εκκρεμούν ζητήματα σχετικά με τη νομική βάση και τον ορισμό της, της ποσόστοσης ε, ενώ ταυτόχρονα η υιοθέτηση της πρότασης ε, θα επιφέρει αλλαγές και στο εταιρικό δίκαιο σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Ε, θα συνεχίσουμε το θέμα, θα πάρουμε την πρόταση της Γαλλίας και της Ιταλίας και θα δουλέψουμε πάνω στην πρόταση της Γαλλίας και της Ιταλίας γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σε διμερείς επαφές με τα κράτη, τα κράτη-μέλη εκείνα που έχουν, μια αρνητική στάση απέναντι στην οδηγία τη συγκεκριμένη. Έχουν ήδη ε, πραγματοποιηθεί κάποιες, ημερές, ε, διμερείς επαφές της υπηρεσίας μας, της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας εδώ στις Βρυξέλλες, με τις κύριες αντιπροσωπείες των χωρών που διαφωνούν, αλλά και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης, προκειμένου ε, να διερευνηθούν οι θέσεις τους όσον αφορά την αντιμετώπιση της υποβληθής σας από τη Γαλλία και Ιταλία πρότασης ως σημείο αφετερίας για το νέο κείμενο της ελληνικής προεδρίας. Αλλά και απ' την άλλη να διαπιστώσουμε μέχρι πού φτάνει η, δια, η διαλλακτικότητα ή η αδιαλλαξία για την ουσιαστική συνέχιση της διαπραγμάτευσης σε περίπτωση πιθανής αλλαγής πλεύσης της Γερμανίας αλλά το, το ότι τοποθετήθηκε μια γυναίκα στο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας νομίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι, όπως ακράδαντα πιστεύω, ότι μια μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως, είναι αυτή η Γερμανία, ε, όπως αυτή είναι η Γερμανία, μια χώρα που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στον νεότερο ευρωπαϊκό πολιτισμό, μια χώρα που έχει για τρίτη φορά ε, γυναίκα πρωθυπουργό, γυναίκα καγκελάριο. Ε, νομίζω ότι αν όλοι μαζί δουλέψουμε ενωμένα, ε, θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε, στο κομμάτι αυτό, με βελτιώσεις οι οποίες θα, θα αποσκοπούν σε, σε μια πιο ακριβή αποτύπωση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σε τρει βασικού άξονε αυτών τη διαδικασία επιλογή των μελών του ΔΣ, των διοικητικών συμβουλίων, το πλαίσιο επιβολή των κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση των χωρών, καθώ και να, διατυπώσουμε μία σαφή, ε, μία σαφή σύνταξη, να έχουμε μία σαφή αποτύπωση της αρχής συμμόρφωση ή επεξήγηση. Ε, όπως είπα, ε, η ελληνική προεδρία ε, είναι σαφώς θετική προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης της οδηγίας αλλά πάντα με, τον σεβασμό, με την ανάγκη σεβασμού των διαφορετικών εθνικών καθεστώτων και συνθήκων και κάτι, μια θέση με την οποία ε, ε έχουμε ξεκινήσει και την επαφή μας με την Επιτροπή. Ε, ελπίζουμε, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Okay. Ε, thank you. Thank you very much and ε, thanks a lot. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε και την παρουσίαση των προθέσεων της Ελληνικής Προεδρίας. Σας ευχόμαστε την πιο επιτυχή δυνατή Προεδρία και παρά το γεγονό ότι τελειώνει η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μαζί σα και πέραν αυτού του χρονικού διαστήματο. Βέβαια είναι δύσκολο αυτό να γίνει την περίοδο των εκλογών, αλλά στο βαθμό του δυνατού θα είμαστε πάντα έτοιμοι να σα βοηθήσουμε. Σα ευχαριστούμε πολύ για την έλευσή σα. για την προσοχή και ελπίζω... Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και ελπίζω να καταφέρουμε να συνεργαστούμε γιατί δεν έχουμε τίποτα διαφορετικό. Όλοι μας, όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δουλεύουν προς την ίδια κατεύθυνση και νομίζω αυτή είναι η υποχρέωσή μας και το χρέος μας. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. då eh, och eh, Να συνεχίσουμε παρακαλώ τη συνεδρίασή μας. Περνάμε στο σημείο 11 σχετικά με τι ανακοινώσει του Πρόεδρου για τις αποφάσεις των ε, συντονιστών. Θα βρείτε ένα κατάλογο ενώπιόν σας ε, και αν δεν υπάρχει αντίρρηση θεωρούμε ότι εγκρίνονται και θα μπουν στα πρακτικά. Και το τελευταίο σημείο για σήμερα είναι το Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διορίσει αντιπροσώπους, διορίζει αντιπροσώπους ε, στο Φόρουμ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και προκειμένου να πληροφορούμαστε, σας καλούμε συχνά εδώ για να μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει εκεί, να μας λέτε τι πηγαίνει καλά, τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικός ο σύνδεσμος αυτός μεταξύ της Επιτροπής μας και του Ινστιτούτου. Επομένως, χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά... Θα τα καταφέρουμε. Τώρα έχουμε εδώ τους κυρίους Ρίκου και την κυρία Λιπρέντη Μαράτου που θα μας εκφράσουν τις εμπειρίες τους και κατόπιν θα έχουμε μια συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Thank you. Ε, ε, dank u voorzitter. in Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να τοποθετηθώ ενώπιον σας. Πριν δύο χρόνια σας είχα ενημερώσει για το τι συνέβαινε στο Ινστιτούτο. Δεν γνώριζα αν πρόκειται να με διορίσετε εκ νέου. Τότε είχα ασκήσει ιδιαίτερη κριτική μέλη του φόρουμ <clears throat> εκεί με έχουν κάπως ε, δώσει κάποιες ε, μικρές επικρίσεις. Και φυσικά όλα τα πράγματα έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, αλλά και οι επικρίσεις μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες. Οι επικρίσεις ε, έγιναν διότι κάποιες χώρες μέλη δεν ήταν παρούσες στο φόρουμ Αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τουλάχιστον τα πάρα πολλοί που παρακολουθούσαν αυτή τη συζήτηση στο φόρουμ μέσω του διαδικτύου. Γιατί αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνονται γνωστές οι απόψεις και οι αποφάσεις για τα δικαιώματα των γυναικών. Εγώ θέλω σας ε, καταπραίνω λοιπόν, δεν θέλω να είμαι ε, σε επίπεδο αντιπαράθεσης. Θέλω απλώς να σας υπενθυμίσω ποια ήταν η άποψη που έχω διατυπώσει ήδη στο παρελθόν και που νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε περαιτέρω πρόοδο. Το IEGE e είναι ένας χώρος που μπορεί να συναθρήσει εμπειρογνώμονες στους τομείς αυτούς. Ακούσατε τα σχόλια της Ελληνίδος Υπουργού. Είναι γεγονός λοιπόν και από αυτά που ακούσαμε ότι όλο και περισσότερο τα πράγματα γίνονται θετικότερα. Αν δούμε τα τελευταία δύο χρόνια, έγιναν πάρα πολλά ε, υπήρξαν πολλές δημοσιεύσεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες. Το κέντρο τεκμηρίωσής μας έχουμε μπορέσει να έχουμε δεδομένα τα οποία έχουμε συλλέξει, τα οποία είναι προσβάσιμα στο κοινό, κρατήσαμε επαφές με τα κράτη-μέλη και για τις δημοσιεύσεις αυτές, πάντα μπορούμε να επιτύχουμε και περαιτέρω πρόοδο. Χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτών οι οποίοι ε, είναι υπεύθυνοι για τις δημοσιεύσεις. Ο στόχος βέβαια δεν είναι η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών, αλλά η συνεργασία. Αυτό το οποίο μπορεί να βελτιωθεί είναι ο ρόλος που διαδραματίζει το ΆΙΓΕ για να παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων που λαμβάνονται. Φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με την εντολή του ΆΙΓΕ, το οποίο δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά πάντα μπορεί να κάνει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δίνει την άποψή του για τα διάφορα τεκθενόμενα το ΑΕΚΕ ως φορέας αλλά δεν μπορεί πάντα να εξασφαλίζει και την απόλυτη ορατότητά του. Το βασικό στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε την πραγματικότητα της ισότητας ανδρών και γυναικών και αυτό είναι φυσικά κάτι το οποίο ενδιαφέρει και την Επιτροπή σας και το Σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε. Με πολιτικές θέσεις, με δηλώσεις, με δημοσίευσεις το θέμα της ισότητας των φύλων είναι ένα εξόχως πολιτικό θέμα και γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εμείς από την πλευρά μας ως ε, αποκεντρωμένος φορέας που δεν έχει ένα πολιτικό ρόλο, αλλά επίσης πρέπει να προωθηθεί και σε άλλους χώρους. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της διαφάνειας εργασίας του ΆΙΓΕ. Φυσικά πρέπει να προσφύγουμε σε εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει πάντα η απαραίτητη ανάδραση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και ημών. Οι δημοσιεύσεις μας, όπως και οι δημοσιεύσεις της Κομισιόν, δίνουν μια εικόνα για αυτά τα οποία γίνονται. Αλλά φυσικά μπορεί κανεί να θέσει το ερώτημα τι κάνουν όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονε. Τι ακριβώς προσφέρουν. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και την διαφάνεια της λειτουργίας του ΑΕΓΕ. Υπάρχει παραδείγματος ένα σεμινάριο το οποίο είχε οργανώσει το ΑΕΓΕ για, την, ε, για το gender mainstream και η έκθεση γι' αυτό έγινε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εμπειρογνώμονες συγγνώμη, και αυτή η έκθεση δεν αναφέρει καν ποια είναι η άποψη του Άγιε. Επίσης το κέντρο τεκμηρίωσης του Άγιε, το οποίο δημιουργήθηκε με σκληρή εργασία για τη συλλογή στοιχείων και τεκμηρίων σε σχέση με την ισότητα των φύλων, Αυτό το κέντρο φυσικά έχει παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι απόλυτα κατανοητό ποια είναι η υποστέμενη αξία που δίδεται από το Άγιε με τη δημιουργία αυτού του κέντρου τεκμηρίωσης. Δεν έχει προσφέρει κάτι καινούριο το Άγιε και νομίζω ότι και εκεί πρέπει να υπάρξει κάποια βελτίωση. Είχα την εντύπωση ότι υπήρξαν πολλές ομάδες ε, προβληματισμού, υπήρξαν ε, ομιλητές οι οποίοι προσκλήθηκαν, υπήρξαν συμπεράσματα από αυτούς οι οποίοι παρακολούθησαν όλα αυτά τα σεμινάρια. Έχουμε Πολλέ στρογγυλέ τράπεζε 10 με 12 άτομα τα οποία συζητούν, θέτουν ερωτήματα, διαφορετικά ερωτήματα σε κάθε τραπέζι, μια σύντομη παρουσίαση στην Ολομέλεια, κάποιο συμπέρασμα το οποίο αντλείται από όλα αυτά. Αλλά αυτά τα συμπεράσματα είναι πολλές φορές λησμονήσιμα ή και λησμονητέα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι σαφές τι προκύπτει από τα συμπεράσματα αυτά και τι μπορεί να κάνει κανείς για όλα αυτά. Νομίζω ότι το σημείο εστίασης πρέπει να είναι και ο δείκτης για την ισότητα των φύλων. Αλλά είμαι κάπως ε, προκατηλημένη σε σχέση με αυτό, γιατί ήμουν και η ίδια πρόεδρος της ομάδας εργασίας που δημιούργησε αυτό το δείκτη. Νομίζω όμως ότι υπάρχει γενική συμφωνία ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε και με εμπειρογνώμες από τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά λοιπόν είναι χρήσιμα για να κατανοούμε βάσει αυτού του δείκτη και τι ακόμα χρειάζεται να γίνει από τα κράτη-μέλη με τη βοήθεια αυτού του στατιστικού στη δείκτη για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο την ισότητα των φύλων. Έρχομαι λοιπόν στο τέλος της ομιλίας μου. Είναι σημαντικό λοιπόν η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η εντολή αυτού του Ιδρύματος, να έχουμε ένα πολιετές πρόγραμμα και στην ε, επαγγελματική μου ζωή Πιστεύω ότι πάντα θα πρέπει να έχουμε ένα πολιετές ε, σχέδιο για να μπορούμε να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Η ομάδα των εμπειρογνωμών, παραδείγματος χάρη, είχε ζητήσει από το Άγγε να πει πέστε μας με την έρευνά σας τι αντιμετώπιση, τι αποτέλεσμα είχε κρίση στην κατάσταση των γυναικών. Εάν οι αρμόδιοι του Άγιε είχαν προβλέψει ότι θα ερχόταν η κρίση, θα μπορούσαν ίσως να έχουν αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προβληματική αυτή. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι το Άγιε μας βοηθάει ιδιαίτερα στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς και το ΜΚΙΟ. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην ε, κυρία Καλησπέρα σα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που με διόρισε ως αναπληρωματικό μέλος ε, στο Ινστιτούτο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Διορίστηκα μόλις τον ε, περασμένο Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 2012 μάλλον, και τον περασμένο Σεπτέμβριο συμμετείχα για πρώτη φορά στο Φόρουμ Εμπειρογνωμών ε, του ΕΙΚΕΙ. Είμαι λοιπόν νεοαφιχτήσα και θα σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις και σημεία που συζητήθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση. Είναι δύσκολο από την πρώτη φορά να σχηματίσει κανείς ε, μία, να πρέπει κανείς σε μία επισκόπηση της, ε, του συνόλου της οργάνωσης του Ινστιτούτου. αναφερθώ σε αυτό που μας δίνει προσθεμένη αξία. Η συνάδελφος έχει μακρά εμπειρία. Έτσι λοιπόν, κατά την τελευταία συνεδρίαση, κατά την τελευταία συνάντηση, το φόρουμ έλαβε χώρα στις νέες εγκαταστάσεις ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό είναι η μόνη ευρωπαϊκή υπηρεσία που ε, βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με την ε, αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και με το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων, είχαμε τις αναφορές στις πρόσφατες εξελίξεις πολιτικής και κατόπιν συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο σημεία. Το πρώτο ήταν ε, η βία ε, με βάση το φύλλο κατά των γυναικών και η εμπειρόγνωμονας ε, παρουσίασε κάποια στοιχεία, καθώς ε, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για τη βία με βάση το φύλλο μεταξύ του 2010 και του 2013. Κατά τη διάρκεια αυτή της περίοδου το Ινστιτούτο έχει συμμετάσχει σε διάφορες πρωτοβουλίες και προετοίμασε μελέτες και εκθέσεις, συνέκρινε διάφορα εργαλεία, βαλιστές πρακτικές, διάφορα δεδομένα επί διάφορων πτυχών ε, της βίας αυτής, όπως είναι ο βιασμός, η οικογενειακή βία, η επίθεση, ο κριτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων, σεξουαλικός καταναγκασμός. Βλέπετε λοιπόν πόσα παραδείγματα έχουμε σεξιστικής βίας. Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε μια μελέτη καινούρια που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πρόκειται για μια μελέτη για τις διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα συλλογής δεδομένων για τη σεξιστική βία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να αναθεωρήσει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που συνεχίζονται με τη σεξιστική βία από τους ευρωπαϊκούς φορείς και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Νομίζω ότι αυτή η μελέτη ε, που υλοποιήθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, έχει ανέβει στο διαδίκτυο. Επίσης, οι πολιτικές στα διάφορα κράτη-μέλη είναι διαφορετικές επειδή υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί και διαφορετικές προσεγγίσεις για τη σεξιστική βία. Αυτό καθιστά την εναρμόνιση και τη συγκριμπότητα των ε, συλλεκτέντων διοικητικών στοιχείων πολύ δύσκολο. Επομένω, το Ινστιτούτο θα μπορούσε να καταβάλει μια προσπάθεια, όπω υπογραμμίστηκε, για να εντατικοποιήσει τη συλλογή των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και να εντάξει πλήρω τα στοιχεία στα συστήματα στα εθνικά συστήματα συλλογή δεδομένων. Επομένω, πρέπει να εστιάσει το Ινστιτούτο καταρχήν στον εργαστή, στον τομέα των κοινών ορισμών, στην ταξινόμηση των συστημάτων, κατηγοροποίηση των συστημάτων και τι μεθοδολογίε και να καθορίσει τι μελλοντικέ ανάγκε ε, και να εναρμονίσει τη συλλογή των δεδομένων. Αυτά είναι ουσιαστικά, αν θέλουμε, να εναρμονίσουμε τη συλλογή των δεδομένων ε, και τις στατιστικές για το φύλλο στην Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα που είχε συμπεριληφθεί στην βερσία διάταξη στην πρόσφατη συνάντηση ήταν η συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το ρόλο των μελών του Ινστιτούτου. Συστάθηκε μία ομάδα εργασία με τρει εβδομάδε που έχει ως στόχο να βελτιώσει την οργάνωση των συναντήσεων του φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να εργαστούν οι εμπειρογνώμονε πιο αποτελεσματικά και φυσικά να ωφεληθεί και το Ινστιτούτο. Προτάθηκε σε προηγούμενε συναντήσει ε, τα εγγραφά να δίνονται από το Ινστιτούτο στα μέλη πριν από την υλοποίηση των συναντήσεων, προκειμένου τα μέλη να μπορούν να έρχονται στι συζητήσει, προετοιμασμένα. Και νομίζω ότι σε οργανωτικό επίπεδο έχει σημειωθεί επαρκή πρόοδος, αλλά φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, η ανάπτυξη της ε, Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για το Φύλλο θα διευκολύνει τη συζήτηση και την επικοινωνία με τα μέλη. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Eurogender Platform, πλατφόρμα, Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για το Φύλλο. Και όπω σα είπε ο Είχαμε και την επίσημη, τα επίσημα εγγένεια, το επίσημο εγγένεια της βιβλιοθήκης, του ΕΙΚΕ και του Κέντρου Τεκμηρίωσης. Είχαμε παρόντες, πολλούς πολιτικούς, εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και ακαδημαϊκούς. Ε, κατόπιν ακολούθησε μία σύνοδος πάνελ για την προσθέμενη αξία του κέντρου τεκμηρίωσης του ΕΕΚΕ για τους ε, χαράκτες πολιτικής, τους ερευνητές ε, και τους ακτιβιστές. Πρόκειται για μια ειδική βιβλιοθήκη και αυτή η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη προ παρέχει πρόσβαση σε περισσότερο από 220.000 πηγές και έχουμε και ένα κέντρο γνώσης για την ισότητα των φύλων. Εκεί έχουμε στατιστικές, μεθόδους, εργαλεία για την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κέντρο τεκμηρίωσης και πηγών, πιστεύω, και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για να παρέχει γνώση σε όλους εμάς. Αυτό για θέματα ισότητας των φύλων. Αυτές είναι οι δικές μου εντυπώσεις, ότι σημειώνεται πρόοδος, η συνεργασία προχωρά σε οργανωτικό επίπεδο και το Ινστιτούτο έχει υλοποιήσει σημαντικές μελέτες και εκθέσεις. Αλλά φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε και περισσότερο τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτο κάνω κάποια σχόλια. Δεν ξέρω αν τα μέλη μας θέλουν να αναλάβουν το λόγο. Σας παρακαλώ, είστε σύντομοι όμως γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πέντε η ώρα έχουμε μία πρόσκληση. Αν δεν θέλετε να με ακούτε να μιλάω σου ειδικά, σας παρακαλώ να κάνετε σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσει να γίνει μια σύντομη απάντηση. Κυρία Μπάουερ πρώτα. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχω την εντύπωση ότι δεν είσαστε τόσο, δεν έχετε τόσο κριτική στάση όπως είχατε το παρελθόν. Την προηγούμενη φορά ήταν πιο έντονη η κριτική σας για ένα μείζον θέμα και είχαμε συμφωνήσει μαζί σας ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα πράγματα. Αλλά είχαμε δει και κάποιες σημαντικές βελτιώσεις εξάλλου στο έργο αυτού του φορέα. Έχετε δίκιο. Βέβαια, ότι το έργο του IG θα μπορούσε να είναι IG, θα μπορούσε να τη χάνει περισσότερο συντονισμού μεταξύ της Κομισιόν ημών και της ε, ΑΕΓΕ και επίσης και άλλων φορέων. Και άλλων φορέων που αντιμετωπίζουν τα θέματα ε, ισότητας των φύλων στον κοινωνικό τομέα. Νιώθω λοιπόν ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι να ζητήσουμε περισσότερες βελτιώσεις υπό τη μορφή καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των φορέων αυτών. Βλέπω να υπάρχει όμως κάποιο κάποιος των θεμάτων, των θεμάτων ισότητας των φίλων στην Κομισιόν. Παλιά ήταν όλα αυτά στην ε, κοινωνική γενική διεύθυνση. Τώρα έχουν περάσει εν μέρει στην κυρία Ρέντινγκ, εν μέρει στην κυρία Μάλμστρομ. Αυτό είναι αντιπαραγωγικό σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συνεργασία και δεν είναι η καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων. Όλα λοιπόν εξαρτάται και από το πώς θα οργανώσουμε καλύτερα το έργο της επόμενης Επιτροπής αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τα, τις απόψεις που μας παρουσιάσατε και θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, συστάσεις σας και στο έργο μας. Ευχαριστώ. Thank you. And, uh, ε, Mrs. Morvai, Morvai, also short, please. Κύριε Μορβάη, εν συντομία. Θα είμαι σύντομη. Όπως ακούσαμε και το πρωί, ο τήσιος προπολογισμό είναι 7,7 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα δαπανίσετε αυτά τα χρήματα, πώς θα τα κατανείμετε και πώς θα ωφεληθούν οι γυναίκες της Ευρώπης σε καιρούς κρίσης. Όταν ακόμη και 7 ευρώ μπορεί να είναι πολύ σημαντικό ποσό. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι λαϊκίζω, αλλά γνωρίζω πώς λειτουργεί ο ακαδημαϊκός χώρος και εγώ ήμουν ερευνήτρια σε γυναικεία θέματα, συμμετείχα σε βιβλία, σε άρθρα, αλλά από τη μια μεριά έχουμε έρευνα που έχει γίνει πολύ σημαντική στην Ευρώπη. Το ποσό που μας αναφέρατε σημαίνει περίπου 300 χιλιάδες ευρώ για κάθε χώρα. Ωραία, πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα ποσά και ποια θα είναι η προσθεμένη αξία της δικής σας δουλειάς, του δικού σας έργου. Πες τι κάνατε, αν μπορώ να ρωτήσω, τι πετύχατε με τα σχετικά ποσά. Κύριε Κορνέλισεν. Δεν ξέρω αν το ερώτημα αφορά τις δύο κυρίες, αλλά ας απαντήσουν όπως νομίζουν. Εντυπωσιάστηκα από την αναφορά της διαφάνειας αφενός και των πολιτικών απόψεων από την άλλη μεριά των ανθρώπων που δουλεύουν για το IGE. Τα αναφέρεται ως ξεχωριστά ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι συνδέονται μεταξύ τους. Πολιτικές απόψεις προφανώς θα έχουν στο FRA. Το ίδιο συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να είσαι στον τομέα αυτόν χωρίς να έχει συγκεκριμένε πολιτικές απόψει, αν δεν πιστεύει σε κάτι και γι' αυτό άλλωστε αφιερώνει και τη ζωή σου στη σχετική έρευνα. Το θέμα είναι όμω η έρευνα από εκεί πέρα να γίνεται αντικειμενικά και αυτό προϋποθέτει διαφάνεια. Συμφωνείτε με την θέση μου αυτή. Και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαφάνειας στον τρόπο επεξεργασία των απόψεων στις ερευνές σας. Και μια ερώτηση μάλλον προς τον Πρόεδρο. Μα συστήσετε να διευρύνουμε την εντολή ώστε να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες ε, περιστάσεις με περισσότερη ευελιξία, εφόσον φυσικά προκύψει αυτή η δυνατότητα. Τι εννοούσατε εφόσον προκύψει, ποια, ποια δυνατότητα. Δεν, δεν, κατάλαβα αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Τι ακριβώς είπατε. Μας είπατε ότι μπορούμε να διευρύνουμε την εντολή του, I, του EIGE, e, έτσι ώστε να είμαστε πιο ευέλικτοι στην αντιμετώπιση των περιστάσεων. Εφόσον προκύψει η ευκαιρία. Θα έχουν τέτοια ευκαιρία. Για ποια ευκαιρία μιλάτε. Εξαιρετική ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Θα τα πω ειδικά όμω ε, από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, δεν ήμουν προετοιμασμένο, αλλά θα το σκεφτώ το ερώτημα. Γενικώ μας επικρίνεται, μάλιστα την περασμένη φορά ήσασταν πιο επικριτικοί ακόμη, τα πράγματα έχουν λίγο ηρεμήσει. Εν πάση περιπτώσει, έχει σημασία η έρευνα να διεξάγεται με διαφάνεια και ειλικρίνεια. Εμεί δεν είμαστε εκεί παρόντε όταν γίνονται οι έρευνε. Προσωπικώ ε, ξέρω ότι έχουμε τακτικέ ε, επαφές πάντως έχει σημασία. Αν κάτι συμβεί, αν κάτι ζήσετε, πρέπει να το μεταφέρετε ως έχει. Ας μην κρυβόμαστε. Αν χρειάζεται να είμαστε επικριτικοί, να είμαστε. Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη πάντοτε. Τώρα στη συμφωνία συνεργασίας που συζητούσαν οι συντονιστές, έχει μεγάλη σημασία να συμμετέχετε στις συνεδριάσεις δύο φορές το χρόνο. Ίσως θα πρέπει να πληθυνθούν οι συνεδριάσεις για να μην υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση από τη μία συνεδρίαση στην άλλη. Τώρα φέτος η χρονιά είναι διαφορετική λόγω εκλογών, όμως καλό θα ήταν να είστε εδώ κάθε έξι μήνες ε, και να μας λέτε τις εμπειρίες σας. Όπως προείπα, τον επόμενο μήνα θα έχουμε τους διευθυντές σας. Ίσως μάλιστα θα ήταν καλό να έρθετε λίγο πιο νωρίς για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν πριν από λίγο. Και να ακούσουμε όχι μόνο τις απαντήσεις, αλλά και τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω τώρα τα τυπικά, τα οργανωτικά, την διαδικασία της συζήτησης ο λόγος σε εσάς. Ε, πολύ γρήγορα όμω γιατί έχουμε μόνο πέντε λεπτά, για το οποίο θα έχουμε και διερμηνία, αλλά όχι περισσότερο. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαπιστώσουμε όλοι μας. Έχω βέβαια δεχτεί επικρίσεις και είπε, είπε σωστά η κυρία Μπάουερ ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμός. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν. Η κυρία Κονέλσεν αναφέρθηκε στην οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Και εδώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα του άρθρου 19 και όχι του άρθρου 2 ένας οργανισμός όπως το IGEM, μαζί με το FRA θα πρέπει να συνεργαστούν και να καταβάλουν προσπάθειες. Είναι διαφορετικές καταστάσεις των γυναικών που είναι ε, ανάπηρες, των γυναικών που είναι λεσβίες, με το ΦΡΑ μαζί θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για όλα αυτά τα θέματα και για τα λεφτά. Θα ήθελα το κοινοβούλιο αυτό να μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο για την ε, ισότητα των φύλων. Και αυτό που ρώτησε η βουλευτής από την Ουγγαρία, πόσο κοστίζει αυτό το Ινστιτούτο για κάθε μέλος του. Δεν νομίζω ότι εγώ είμαι αυτή η οποία πρέπει να κρίνει τα οικονομικά θέματα. Αυτό μπορείτε να το θέσετε το ερώτημα στην ε, Γενική Διευθύντρια του ΆΙΓΕ όταν πρόκειται για θέματα προϋπολογισμού. Θα πρέπει να ξαναδούμε λοιπόν και τον κανονισμό για το Ίδρυμα αυτό. Είναι 5-6 χρόνια που έχει δημιουργηθεί αυτό το Ινστιτούτο και υπάρχει βέβαια και ο κανονισμός ο οποίος προβλέπει να γίνει κάποια βελτίωση μετά από μια ενδιάμεση περίοδο για τον κανονισμό του Ιδρύματος. Αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λάβει κανείς και υπόψη το κατά πόσο θα πρέπει να ενισχυθεί και η εργασία του οργάνου αυτού. Και το θέμα της ε, διαφάνειας που νομίζω και αυτό το έθιξε η κυρία Κονέλσεν, Όταν αντιμετωπίζει κανείς με την, τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην ε, κοινωνία, προφανώς πρέπει να μπει και στην πολιτική προβληματική. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας αποκεντρωμένος φορέας. Θα πρέπει να ζήσουμε με αυτή την αντίφαση όμως. Γι' αυτό σας λέω ότι οι συνεργάτες του άγε, προσπαθούν να αφήσουν στο περιθώριο τις πολιτικές τους απόψεις που δεν είναι πάντα εύκολο. Τώρα, ε, όπως είπε και η κυρία Βιλερμίν ε, και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, υπάρχει ένας κατακαιρματισμός των θεμάτων και ίσως επαναλαμβάνονται θέματα μελετών που κάνει η Κομισιόν και από το ΕΓΚΕ, δηλαδή και συχνά βλέπω ότι δεν χρησιμοποιούνται πολύ στα reports εδώ του Κοινοβουλίου, χρησιμοποιείται τα, τα δεδομένα από το ΕΓΚΕ, το, τον συνθετικό δίκτυο ισότητας. Όλα αυτά είναι δουλειά βέβαια ε, που έχει γίνει και έχει παραχθεί και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν αυτά τα, τα δεδομένα και οι στατιστικές αναλύσεις. Όπως ελέγχθηκε κατά τη τελευταία συνάντηση, θα εντατικοποιήσει την συνεργασία με τη Eurostat το ΕΙΓΕ ώστε να μπορέσει να ε, παράξει καλύτερες στατιστικές πιο αξιόπιστες για να έχουμε για τη θέση της γυναίκας. Ε, ε, στο ερώτημα ότι τι παράγει το ΕΙΓΕ και, γιατί, τι, ποιο είναι το όφελος για τις γυναίκες της Ευρώπης νομίζω ότι το ότι υποστηρίζει τις προεδρίες ότι κάθε έξι μήνες κάνει μια διαφορετική μελέτη στα πλαίσια της, του, του Πεκίνου, της πλατφόρμας του Πεκίνου, ένα από τα 12 αυτά θέματα που ήταν η φτώχεια, η οικονομία, η υγεία των γυναικών και όλα αυτά και διερευνάτε σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικό για να γνωρίζουμε τι γίνεται για αυτά τα ζητήματα. Είναι πανευρωπαϊκές έρευνες, δεν αφορούν μόνο μία χώρα, γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης το ότι ε, παρατίθενται συστάσεις, ε, προτάσεις, ε, καλές πρακτικές και όλα αυτά είναι που συσσωρεύεται μία γνώση η οποία μπορεί να μας χρησιμεύσει μετά στις πολιτικές, στο νόμο, γιατί νομοθετεί εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν βέβαια, με πρωτοβουλίες της Κομισιόν. Οπότε όλα αυτά, η συσσωρευμένη γνώση νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Τα ζητήματα διαφάνειας και μεθοδολογίας βέβαια είναι αρκετά πολύπλοκα. Θα πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα και να ξέρουμε καλύτερα πώς διεξάγονται οι μελέτες και πώς ε, αυτά τα δεδομένα τα οποία ε, γίνονται σύνθετες αναλύσεις αν τελικά ε, τα συμπεράσματα και οι τάσεις που δείχνουν είναι αξιόπιστες. Ε, να υπάρχει δηλαδή και μια αξιολόγηση αυτών των δεδομένων γιατί είναι, πραγματικά είναι ειδικότερα ο δείκτης ισότητας θα πρέπει να αποτυπώνει τις τάσεις της Ευρώπης και των χωρών ειδικότερα. νομίζω ότι είναι ένα ακαδημαϊκό ακαδημαϊκό κέντρο έρευνας το οποίο πολλές φορές διαρωτόμαστε τι παράγει ένα ακαδημαϊκό κέντρο έρευνας παράγει γνώση. Δεν μπορούμε να, ούτε να δώσουμε άλλα προϊόντα γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει να μπορέσει να βελτιωθεί ώστε να είναι καλύτερη η απόδοσή του και πιο οργανωμένες οι συναντήσεις του expert forum. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρουσιάζετε εδώ τις ε, απόψεις σας από το φόρουμ και ελπίζω να μπορείτε να ξανάρθετε. Και έτσι όπως έχουμε συμφωνήσει, αυτό γίνεται δύο φορές το χρόνο. Ίσως να μην τα καταφέρουμε φέτος, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε τακτική επαφή και να λαμβάνουμε πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο Ινστιτούτο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που περιβρεθήκατε και ολοκληρώνουμε εδώ τη σημερινή συνεδρίαση. Ζητώ συγγνώμη από τις διερμηνείς που καθυστερήσαμε λίγο, αλλά θα επαναρθώ στην επόμενη φορά, λέει ο Πρόεδρος.